Good morning, ladies and gentlemen. I think we Θα ξεκινήσουμε. Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Ξεκινώντας, να μου επιτρέψετε να σας ευχηθώ καλή χρονιά να σας ευχηθώ ένα 2019 γεμάτο ευτυχία και υγεία. Ελπίζω όλοι να πετύχετε αυτή τη χρονιά τους στόχους που έχετε θέσει. Καλή σας τύχη. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση λοιπόν, την έκτακτη αυτή συνεδρίαση, η υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν σχόλια. Έγκριση των προηγούμενων πρακτικών. 25 Οκτωβρίου, 15 Νοεμβρίου και 21 και 22 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα online ως συνήθως και αν δεν υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσης συνεδρίασης θα θεωρηθούν δεκτά. στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω μία να κάνω, πολύ σύντομη. Για την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη Τρίτη, ε, θα έχουμε την πιο σημαντική ψηφοφορία νομίζω αυτής της ε, περίοδου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό των κοινών προβλέψεων. Θα το ολοκληρώσουμε στις 22 το πρωί. Είναι δυνατόν να γίνει. Υπάρχουν άνω των 100 τροπολογιών συμβιβαστικών. Οι εισηγητές είναι ήδη προπαρασκευασμένοι. Έχουν ενημερώσει και τους σκιώδεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Θα χρειαστούμε το σύνολο του πρωινού την Τρίτη το πρωί, την Τρίτη το απόγευμα θα ακούσουμε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας και θα ανταλλάξουμε απόψη μας με την Επίτροπο το τέλος του απογεύματος θα ακολουθήσει μια δεξίωση, μια μικρή δεξίωση. Το αξίζουμε μετά από τη δύσκολη δουλειά που κάναμε για τον κοινό κανονισμό. Νομίζω ότι αξίζει να πιούμε κάτι μαζί. Λοιπόν, αυτό να είμαστε πειθαρχικοί λίγο σε σχέση με το χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες για την χρηματοδότηση της διαχείρισης και της εποπτείας της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ο κύριος Μπόγκοβετς, θέλετε κάτι το εισαγωγικό να πείτε? Όχι, οπότε περνάμε απευθείας λοιπόν στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν με την πρώτη. Για την τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 50. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία και εδώ. Δεκτή. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή από κοινού 11 και 27 ψηφίζεται η κατά αποχές δεκτές 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 και 14 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή από κοινού 54 και 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές, 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 55 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 56 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, από κοινού 59 και 60 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογίες τώρα 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή από κοινού την 65, την 66, την 68, την 85 και την 86 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 70, 71, 72, 73, 74 από κοινού υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Από 70 μέχρι και 74, αν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 και 78 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 και 80 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. 81 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 81 ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 82. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογίες 97 μέχρι 106 ε, μια μεγάλη ομάδα τροπολογιών ψηφίζονται από κοινού Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα τροπολογία 108, 109, 110 και 111 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή ομάδα τώρα τροπολογιών από 32, 33, 34, 35 και 36 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές, 120 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 121 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 123 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 37 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1 και 38 από κοινού. Υπέρ, κατά αποχές δεκτές 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή από κοινού τώρα την 42, την 57, 58. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Από κοινού την 43 και την 69 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48, 49 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο με ηλεκτρονική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί έχετε ένα μέλος επιπλέον. Ε, έγινε ένα λάθος από τους υπολογιστές. Καλώς λοιπόν, 34 ψηφίζουν, οπότε είναι σωστό. Γίνεται δεκτή η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπόγκοβιτς. Καλώς. Συνεχίζουμε. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ο τίτλος είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Πρόκειται για γνωμοδότηση που ετοίμασε για μας ο κύριος Ομαρζέ όσον αφορά την γεωργική πολιτική. Θέλετε το λόγο κύριο Μαρζέ? Όχι. Ωραία. Είναι πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση κανονισμών κλπ. κλπ. Έχετε όλα τα νούμερα, τις ονομασίες κτλ. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω τον τίτλο. Ε, είναι πιο μεγάλος ο τίτλος από τον ίδιο τον κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν, αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμός 20. 20, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 21. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. τροπολογίες 22 και 23 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 22 και 23. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τώρα, τροπολογία αριθμός 1, 2 και 3. Μαζί ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογίες 24, μόνο 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αν θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και 25 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογίες 8 και 26 που είναι ίδιες, τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και τροπολογίες 9 και 27 μαζί για την ίδια υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 καταπίπτει συνεπώ. και τώρα ψηφίζουμε για την 11 και 29 που είναι ίδιε, μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 12 και 30 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριο Μερζέ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα, επόμενη ψηφοφορία είναι η γνωμοδότησή μας που ετοίμασε η κυρία Μαλετίτς για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Θέλετε να πείτε κάτι προηγουμένως κυρία Μαλετίτς, όχι. Οπότε ψηφίζουμε. Και αρχίζουμε με την τροπολογία 68. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70. Υπέρ, α, χωριστή ψηφοφορία στην 70. Κατά τμήματα, μάλλον, κατά τμήματα. Αλλά δεν το έχω εγώ εδώ, λέει πρόεδρος. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Για την τροπολογία 70 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 και 78 που είναι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 84. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 85. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 Έχουμε την 93, αλλά διαβάζετε το μήνυμα. Έτσι, 94. Υπέρ, λέει πρόεδρος. Α, πρώτο τμήμα. Ναι, είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, έκανα λάθος, λέει η πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 93. Συγγνώμη γι' αυτό. 93 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ της 99, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 106. Όπως και 107 και 108 και 109 είναι η ίδια ιδέα από ό,τι φαίνεται. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 111. Όχι, πάμε κατευθείαν στην 11, στην τροπολογία 11, επειδή απορρίφθηκαν ακριβώς. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 130 και 131 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε με τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Δεν την ψηφίζουμε και πάμε στη συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25. Ε, όχι, 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 26. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Απορρίπτεται. Μία ψήφος παραπάνω. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 δύο τμήματα. Με την προφορική τροπολόγηση. Έχει κανείς αντίρρηση για την προφορική τροπολόγηση πρώτο τμήμα της 55 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά οχές, δεκτή. Δεν ψηφίζουμε την 58, 59 υπέρ κατά οχές, απορρίπτεται. 60 με προφορική τροπολόγηση υπάρχουν αντιρρήσεις όχι. 60 με την προφορική τροπολόγηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 και 61 ταυτόσιμε υπέρ κατά αποχές Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος Τις 64 Άρχεται. Πέρας. Με συγχωρείτε δεκτή. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ονομαστική άρχεται. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μάλετ. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Θέσπιση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Έχουμε γνωμοδότηση. Ο συντάκτης είναι ο κύριος Τσέλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις φράσεις. Πρώτον, τα διαθροτικά ταμεία και οι κανονισμοί που ισχύουν μπορούν να συνδυαστούν με τα μέσα της πολιτικής γειτονίας και προενταξιακής βοήθειας. Αυτό που πρέπει να διαπιστώσουμε στις συζητήσεις ε, που έκανα στις χώρες αυτές αλλά και με εκπροσώπους ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών από τις ε, χώρες προσένταξη και τις χώρες γειτονίας είναι ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι τώρα στο σύστημα της προσέγγισης των χωρών αυτών προς την Ένωση. Και γι' αυτό έριξα ιδιαίτερο βάρος σύμφωνα και με την Επιτροπή Περιφερειών έριξα βάρος στο να καλέσουμε την Κομισιόν να συνεργάζεται περισσότερο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και φορείς. Και θα ήθελα να συμφωνήσετε συνάδελφοι σε αυτό. Και επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τους κοιόδης και τα μέλη της γραμματείας που βοήθησαν την εκπόνηση αυτής της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ψηφίσουμε λοιπόν αυτή την γνωμοδότηση 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές έλεγχος τη 48 άρχεται Πέρας. Δεκτή, λέει η πρόεδρο Α, όχι, α, απορρίπτεται. Μία ψήφος παραπάνω Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται πιστεύω, αλλά έλεγχος. Της 71. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Μία θετική ψήφος παραπάνω. Οπότε η 72 καταπίπτει, 73 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15, ε, 79, λέει πρόεδρος, υπέρ κατά. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, 15. Mm. Συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα με το κατάλογο ψηφοφορίων που έχω μπροστά μου. Α, ωραία. Ωραία. 15 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 79 τώρα. Υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. 80 υπέρ κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Α, συγγνώμη. Συμβαστική δύο, όπως έλεγα λοιπόν, υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 26. Υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 28. Υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 29. Υπέρ κατά αποχές, Απορρίπτεται. Η 30 έχει αποσύρθει. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή πιστεύω. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και συγχαίρουμε τον κύριο Τσέλα. Ευχαριστώ πολύ γιατί τα πήγαμε πολύ καλά. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες σε λιγότερο από μία ώρα. We continue now with Και τώρα θα περάσουμε Can we, can we continue? Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με την εξέταση του σχέδιου γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Για το 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ετήσια ε, έκθεσή της τον, τον Νοέμβριο. Η επισκόπηση αυτή είναι το κύριο όργανο για να εξηγήσει ποιε είναι οι οικονομικέ και κοινωνικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη ε, χρονιά. Επίση, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τον ε, τήσιο κύκλο συντονισμού τη οικονομική πολιτική, όπου οι εθνικέ πολιτικέ εξετάζονται σε ενωσιακό επίπεδο. Η ΕΚΟΝ είναι η αρμόδια επιτροπή, συντάσσει μία έκθεση για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη και η Ρέτζη αποφάσισε να κάνει μια γνωμοδότηση. Είμαι η εισηγήτρια και σήμερα παρουσιάζω το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Οπότε θα πάρω και το λόγο για να την παρουσιάσω. Και κατόπιν θα προτείνω και προθεσμία για τις τροπολογίες. Λοιπόν, το σχέδιο γνωμοδότηση για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη για το 2019. Όπως ξέρετε, είναι βασικό στοιχείο που ε, καθορίζει τον, ε, την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το επόμενο έτος. Τα κύρια σημεία που αναφέρει η γνωμοδότηση για το 2019 Α, είναι τα εξή. Η οικονομία της Ένωσης εξακολουθεί να αναπτύσσεται, έχει αυξηθεί πολλή απασχόληση, αλλά παρόλα αυτά ο αριθμός των ε, σημείων ε, όπου είμαστε ακόμη ευάλωτοι αποδεικνύει ότι δεν έχουμε ακόμη βοηθήσει τους πάντες. Συγγνώμη, γνώμη συμφωνεί με την άποψη ότι οι επενδύσεις, οι καινοτομίες, η γνώση και οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις είναι το κυριότερο για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συνεκτική και τονίζει ότι οι επενδύσεις ε, ε, με βάση την πολιτική συνοχή μαζί με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις παίζουν τεράστιο ρόλο για να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη η συμπερίληψη όλων και οι δυνατότητε τη διοίκηση και των θεσμών. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν και περαιτέρω μέτρα για να μοχλεύσουν τι δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει, για να βελτιστοποιήσουν την προστιθέμενη αξία των πόρων τη ε, πολιτική συνοχή και την ε, ε, συνέργειά τους και συμπληρωματικότητα με τα άλλα οικονομικά μέσα της Ένωσης. Η γνωμοδότηση καλωσορίζει την πρόταση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και του ε, στενού δεσμού μεταξύ της πολιτικής συνοχή και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η γνωμοδότηση καλωσορίζει επίσης την ισχυρότερη εστίαση του οικονομικού εξαμήνου για το 2019 στι ανάγκε επενδύσεων που πρέπει να είναι η βάση για τι προγραμματικέ αποφάσει για την περιοδο 2021 2021-2027. Και έχουμε ένα νέο παράρτημα που προτείνουμε στις ε, αναχώρα εκθέσεις του 2019. Σε αυτό το παράρτημα θα πρέπει να αναφέρονται οι ανάγκες επενδύσεων με βάση το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Αυτές ε, πρέπει να εντοπιστούν λοιπόν, αυτές οι ανάγκες. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω απλούστευση και περισσότερη ευελιξία μεταξύ των ταμείων, προγραμμάτων και μέσων τη Ένωση, ούτω ώστε η χρηματοδότηση να γίνει απλούστερη, απλούστερη και πιο αποτελεσματική. Αυτή είναι η σύντομη παρουσίαση της γνωμοδότησής μου. Και τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδης για αυτή την γνωμοδότηση. Πρώτος είναι ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε αυτή την γνωμοδότηση, η οποία είναι σύντομη Όλα αυτά θα έλεγα ότι περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία. Και εγώ θα είμαι σύντομο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το αισιόδοξο πνεύμα της παρουσίασης και του περιεχομένου. Είναι θετικό να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά την σημασία που έχει η πολιτική συνοχή. Αν δεν το κάνουμε εμείς δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και από πλευρά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 κάτι το οποίο θα αυξήσει ουσιαστικά και τα έσοδά τη. Φύτο. Συμφωνούμε με τη γνωμοδότησή σας, συμφωνούμε και με τον Βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις του Brexit στην πολιτική συνοχής. Εμείς θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πάντως στα θέματα της πολιτικής συνοχής και του Brexit. Ευχαριστώ. Πολύ. Γνωρίζετε τις θέσεις της ομάδας μας. Είμαστε κατά της ε, έγκρισης αυτής για το σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που επιδεινώνει την κατάσταση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς ε, υιοθετούμε μια θέση που είναι συνεπής προς τις συνήθειες τοποθετήσεις μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την ε, Πρόεδρο για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει για να καταλήξει σε αυτή την πρόταση και ευχαριστώ και όλους τους συναδέρφους που συμμετείχαν στο έργο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ανάπτυξη το 2019 θα είναι αυτή που είναι. Οι προβλέψεις βέβαια μπορεί να μην επαληθευτούν. Το 2019 θα έχουμε πολύ μεγάλη στήριξη σε σχέση με την περίοδο 2014-2021. Το 2014 μόνο το 20% των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν, ενώ το 2019 ε, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω 30%. Το πραγματικό ποσό της στήριξης δεν θα είναι όμως αντίστοιχο γιατί όσο πιο πολλά έργα αναθέτεις, τόσο πιο ακριβά γίνονται. Ελπίζω ότι στην επόμενη περίοδο, 21 με 27, θα μπορέσουμε να έχουμε μια κατανομή πιο ισόρροπη των επενδύσεων. Οι χώρες εκείνες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες εξαρτώνται πάρα πολύ από την ευρωπαϊκή στήριξη, από τα διαρθρωτικά και άλλα ταμεία. Το βλέπουμε ότι όταν ε, μια χώρα στο τέλος της περίοδου ε, παίρνει κάποια χρηματοδότηση, στην αρχή της επόμενης περίοδου υπάρχει μεγάλη μείωση. Και υπάρχει μια άνηση ε, κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη στις περιφερειακές περιοχές. Οι πρωτεύουσες αναπτύσσονται πιο γρήγορα, η περιφέρεια όμως πιο αργά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, ώστε οι χώρες μέλη να διασφαλίσουν μια συνολική και ισότιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτεια. Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε και το εξής. Οι χώρες εκείνες οι οποίες ε, σήμερα ε, χωρίζονται σε μικρές περιφέρειες Παλιά ήταν μια περιφέρεια, εδώ τώρα έχουν μια διαφορετική διοικητική δομή. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάπτυξη ε, πρέπει να είναι πιο ισότιμη μεταξύ των περιφερειών. Και όταν μιλάμε για το Ταμείο Συνοχής ή για άλλα χρηματοδοτικά μέσα, είναι πολύ σημαντικό ο δικαιούχος να νιώσει τα ωφέλη από το ταμείο αυτό, όχι μόνο οι οργανωτές, οι διαχειριστές των κονδυλίων. Είναι σημαντικό να υπάρχει πιο στενή σύνδεση με την πολιτική συνοχής. Μερικές φορές το χάσμα μεταξύ των διάφορων περιοχών μπορεί να αυξηθεί. Και θέλω να το τονίσω ότι από την αρχή του 2021 Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις της Κομισιόν, χρήματα από τη συνοχή και τα διορθωτικά ταμεία θα μειωθούν σημαντικά. Γι' αυτό και είναι ζωτική σημασία για το 2021 και το 2022 οι χώρες μέλη και ίσως και η Επιτροπή να πρέπει να αναθεωρήσουν τα προγράμματα για να μην υπάρχουν υπερβολικές δαπάνες σήμερα, χωρίς ε, απτές επιπτώσεις. Γιατί έτσι θα επηρεαστεί συνολικά η ανάπτυξη όταν θα μειωθεί η χρηματοδότηση. Και υπάρχει και το Brexit βέβαια που και αυτό θα έχει επιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Κυρία Δεμάτο. Σύντομα θα ήθελα να εκφράσω τη δική μας θέση Είμαστε κατά τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ακόμα και ο Γιούγκερ κατανόησε ότι η λιτότητα κάνει περισσότερες, προκαλεί περισσότερες βλάβες παρά ωφέλη αλλά στα πλαίσια ενός συμβιβαστικού πνεύματος θα προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε τουλάχιστον την πολιτική συνοχή, η οποία έχει άλλους στόχους, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ε, λιγότερο ε, αναπτυγμένες περιοχές και Δυστυχώς από ό,τι λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαφορά ανάμεσα στις πλούσιες και στις φτωχές περιοχές θα παραμείνει υψηλή. Πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ευχαριστούμε άλλος κανείς από τη Ρέτζη για αυτό το θέμα. Όχι. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τώρα. Είναι η κυρία Παρβάρα Βαλεντίνοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη μίλησατε για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. Θα ασχοληθώ με τι καινοτομίε που θα κάνουμε το 2019. Ο κύκλο που ξεκινάει το 2019 είναι εν μέσω διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου θα ληφθούν αποφάσει για τι δημόσιε επενδύσει για αρκετά χρόνια. Οι επενδύσει συνέονται ε, στενά με τι διαστατικέ μεταρρυθμίσει. Οι επενδύσεις ε, δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές δημιουργούν καλύτερο κλίμα για τις επενδύσεις. Όλες οι πολιτικές πρέπει να είναι συμπληρωματικές και θα βοηθηθούν και οι δύο διαδικασίες. Γι' αυτό στον κύκλο αυτό θα ασχοληθούν περισσότερο με την αποτίμηση των αναγκών επενδύσεων, ούτως ώστε οι αποφάσεις προγραμματισμού για την περίοδο 2021-2027 να γίνουν με καλύτερο τρόπο. Στι εκθέσει του 2019 που θα υποβληθούν το Φεβρουάριο, εξετάζουμε τι ανάγκε επενδύσεων σε κάθε χώρα. Και όπου έχει έννοια και την περιφερειακή και κλαδική διάσταση. Με βάση αυτέ τι αναλύσει θα υπάρξει ένα νέο παράρτημα που θα καθορίζει αυτέ τι ανάγκε και τι σημασία έχουν για το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και το Ταμείο συνοχή για την επόμενη περίοδο. Έτσι θα έχουμε μια καλή βάση για το διάλογο με τα κράτη-μέλη. Με βάση τις εκθέσεις αυτές θα εντοπίσουμε στις, προτάσει στις προτάσεις μας για τις αναχώρα ε, συστάσεις τους τομείς προτεραιότητας για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Αυτά τα νέα στοιχεία όμως δεν ε, αλλάζουν ε, τον κύριο στόχο που είναι το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να γίνουν οι σωστές διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις. Και είναι ουσιώδες ε, να στερνιστούν οι χώρες την ανάγκη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό έχουμε διμερείς ε, συναντήσεις με τα κράτη-μέλη για τα θέματα που αφορούν κάθε χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ω εισηγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση, συντάκτρια, Ευχαριστώ πολύ όλους τους Κιώδης. Θα είναι πολύ σημαντική συμβολή μας για να καταδειχθεί ο ρόλος της πολιτικής συνοχής. Και τα θέματα που θα επηρεαστούν από το Brexit. Πώς θα επηρεαστούν οι αιρεσιμότητες και η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των κρατών μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τις τροπολογίες. Τρίτη 22 Ιανουαρίου, 18 η ώρα. Είναι την επόμενη Τρίτη. Αλλά πρέπει να είναι τόσο σύντομη η προθεσμία λόγω του χρονοδιαγράμματος εργασιών της ΕΚΟΝ. Λοιπόν, τέλος της ημέρας, επόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα με τα, με τα διάφορα. Υπάρχουν διάφορα. Λοιπόν, υπενθυμίζω, η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει την 3η 22 Ιανουαρίου το πρωί και το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ωραία, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Σα ευχαριστώ πολύ.